ότι ο κύριος Μίχαηλ Τουξάνου εξελέγει από τις 2 Μαρτίου 2015, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κύριο Εντουάρ Ραούλ Χέλβικ. Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές με ενημέρωσαν ότι η κυρία Εστεφάνια Τόρες Μαρτίνες εξελέγει από τις 20 Μαρτίου. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αντικαταστήσει τον κύριο Πάμπλο Ετσενίκε Ρόμπα. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη την εκλογή αυτών των δύο συναδέλφων. Τους ε, καλωσορίζω και τους υπενθυμίζω ότι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεδρίασε 23 Μαρτίου